Ευχαριστώ πολύ. Γραπτή δήλωση 61 του 2010 υποβληθήσα από τους συναδέλφους Τόμσεν, Λίνε, Φιγκερέιδο, Ντέλη και Πρώτα Ζιέβιτς. Ο κύριος Ντέλη έχει ζητήσει το λόγο. Πρόκειται για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αστέγους. Ε, σύμφωνα με τον κανονισμό 123 ε, θα μεταδοθεί και θα δημοσιευθεί στα κείμενα της ε, προηγούμενης Ολομέλειας. Για 30 λεπτά Καρίμα Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη συγκίνηση εξ ονόματος των συναδέλφων Τόμσεν, Λίνεφ, Γκυρέιδο και Πρότασιεβίτσε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την στήριξη ε, που δώσατε στην δήλωση 61-2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην ε, εμβληματική της πρωτοβουλία παρουσιάζει μια πλατφόρμα για τους άστεγους. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να ξεχάσουμε τα ωραία λόγια. Πρέπει να περάσουμε στις πράξεις. Συγκεκριμένες προτάσεις προτάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε το 2015 κανένας άστεγος πια να μην κοιμάται στους δρόμους. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένες γιορτές και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Μπεσέ εξ ονόματος των τριών συναδέλφους ε, μου Πετικάνεν, ε, Σαρμπού και Ντέιβις ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 410 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπέγραψαν την γραπτή δήλωση 71-2010 έτσι ώστε να ζητήσουμε ενίσχυση της προστασίας των καρχαριοειδών. Πρόκειται για ένα είδος ε, το οποίο ε, κατακρεουργείται στην θάλασσα ε, κυρίως μέσω της αποκοπής των πτερυγίων τους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που υπερψηφίσατε δηλαδή που υπογράψατε συλλογικά αυτήν την δήλωση ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την προστασία του είδους αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ε, πρόκειται για πολυπληθείς ψηφοφορίες. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και βάσει της απλουστευμένης διαδικασίας